Denis Dormula. Ah Καλημέρα συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη, ο πρόεδρος Κλοντ Μωράης δεν μπορεί να είναι σήμερα στην συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας γιατί έχει ένα μικρό πρόβλημα υγείας έχουμε την εξή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 7.1 παρουσίαση της κατάστασης εξέλιξης του τριμερούς διαλόγου σχετικά με την οδηγία για τις ποινικέ διαδικασίες όσον αφορά το τεκμήριο αθωότητας και την παράσταση στην δίκη. Ε, το σημείο 5, ανταλλαγή υπόψεων ε, για το θέμα της Τουρκίας ε, και της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ρούτα θα πάει σήμερα στην Τουρκία και θα μας ε, πει στην επόμενη συνεδρίασή μας διάφορα πράγματα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα το σημείο για τον προϋπολογισμό επίσης πρέπει να το αφήσουμε γιατί ο κύριος Νίτερ Μουλέρ είχε κάποιο πρόβλημα με την πτήση του. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αντίρρηση, ε, ε, γκρίνουμε την ε, ημερήσια διάταξη με αυτές τις τροποποίησεις. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίρρηση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η διερμηνία στα κροατικά και... και στα γοηδελικά δεν υπάρχει σήμερα. έχουμε Επίσης το θέμα του καθορισμού των ε, συντονιστών. Η κυρία Μουσολίνη είναι η συγγήτρια για την συνεργασία, ε, τη στρατηγική συνεργασία όσον αφορά ε, την μάχη κατά της τρομοκρατίας μεταξύ των αραβικών χωρών και, του, και της Γιουροπόλου, Ο κύριος Φοντάνα είναι ο εισηγητής ε, για την έκθεση σχετικά με την στρατηγική συνεργασία μεταξύ ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, και της Europol μετά από την αλλαγή ομάδας της κυρίας Μακοβέη που πήγε τώρα στο ECR το θέμα στο οποίο ήταν η συγγήτρια ή η σκιώδης τα θέματα αυτά ε, άλλαξαν εισηγητή. Η κυρία Νενοβέ είναι υπεύθυνη για τον κανονισμό σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τρίτο σημείο τώρα. Εγκρίνεται τη συστάση των συντονιστών σύμφωνα με το άρθρο 205 του κανονισμού. Ωραία. Ένα σημείο... Ένα... Το Σεπτέμβριο του 2015 η Κορεπέρ άλλαξε την έκθεση που εγκρίθηκε σχετικά με την απλοποιημένη διαδικασία για την τροποποίηση του άρθρου 52 του ε, κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής ΛΥΒΑ για τις εξής προτάσεις της Επιτροπής. Πρώτον, πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ε, που ε, συντομεύει κάποιες ε, ε, διατάξεις για τον χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης Επίσης, διάφορες πράξεις σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στα ποινικά ζητήματα. Μια άλλη πρόταση σχετικά με την συνεργασία, την αστυνομική και την νομική για ποινικά ζητήματα. Και για τα τρία ζητήματα αυτά θα είναι η συγκητής ο Κλόντ Μωράης και η ψηφοφορία θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου του 2015. Πέμπτη στις 3 θα γίνει ε, η ψηφοφορία να έχετε μαζί σας ε, τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τώρα πάμε στο σημείο 4 παρουσίαση της κυρίας Μαρτασικά ε, γενική στρατηγική διευθύντρια για από την DG Home, Strategy General Affairs. Ε, ο κύριος Ρέτε δεν μπορεί να είναι στην ε, συνάντησή μας σήμερα, θα είναι στην Τουρκία και γι' αυτό δίνω το λόγο στην κυρία Σιγκάν, η οποία ήδη έχει συμμετάσχει στην συνάντηση των συντονιστών και έχει το λόγο. Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ ε, για το γεγονός ότι δώσατε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να συζητήσει την κατάσταση εφαρμογής ε, του, ε, της Ευρωπαϊκής Ατζέντας ε, για την μετανάστευση και να επανέλθει σε εσά. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Πάντοτε ξεκινάμε λοιπόν με αυτά τα γενικά νούμερα των αφήξεων από τον Ιανουάριο του 2015 αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 750.000. Από τότε που εγκρίθηκε η ατζέντα για την ε, μετανάστευση στα μέσα του Μαΐου, έχουμε συνεργαστεί για μια συντονισμένη απάντηση στην κρίση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω κάποια ενημέρωση σχετικά με τα επιτεύγματα που έχουν ε, υπάρξει με βάση την ατζέντα. Θα μιλήσω για την ίδια την κρίση. Καταρχάς να μιλήσω για το γεωπολιτικό υπόβαθρο που στην ουσία ε, είναι και η πηγή αυτής της τρέχουσας η κατάσταση στη Συρία και στη Λιβύα δεν πρόκειται να βελτιωθεί από ό,τι φαίνεται στο προσοχές μέλλον και αυτό σημαίνει ότι η κρίση δεν είναι πρόσθεσμη, δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη, έκτακτο περιστατικό και ο εκτοπισμός των ε, πληθυσμών λόγω της κατάστασης στη Συρία θα συνεχίσει. Επίσης θα αυξηθεί και η ε, ροή από το Αφγανιστάν λόγω της κατάστασης που βρίσκεται ακόμα σε ε, δύσκολη θέση. Τον Ιούνιο είχαμε την ε, κορύφωση ε, των αφήξεων, οι οποίες κάπως μειώθηκαν τον Αύγουστο από την Αφρική, Ερυθρέα, Νιγηρία, Σομαλία και Σουδάν είναι οι χώρες προέλευσης. Η Σύνοδος Κορυφής της Βαλέτα που ξεκινά αύριο, είμαι πεπισμένη ότι θα μπορέσει μέσα σε ένα διήμερο να δώσει την κατάλληλη απάντηση και τα απτά αποτελέσματα που θα ενισχύσουν τη συνεργασία μας με τις αφρικανικές χώρες. Αυτή η σύνοδος κορυφής είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τη σχέση μας με τις αφρικανικές χώρες και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι απλώς η αρχή. Έχουμε μια σειρά επαφών με τους Αφρικανούς εταίρους μας βάσει διμερών, περιφερειακών και άλλων ε, διαδικασιών. Περιφερειακές είναι η διαδικασία του Ραμπάτ και του Χαρτούμ, αλλά δεν έχουμε πραγματικά ξεκινήσει από το μηδέν, υπάρχει υπόβαθρο και νομίζω ότι αυτό θα αποδώσει. Υπάρχει και το πνεύμα συνεργασίας με τους εταίρους μας που ε, δείχνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα project ε, που μπορούν να εφαρμοστούν από κοινού, από κοινού τους επόμενους μήνες. Ε, επίσης, πρόσφατα είδαμε αλλαγή της αιστείας της κρίσης προς τα ανατολικά αυτή η οδός τώρα ε, βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Στην απάντησή της λοιπόν η Κομισιόν έχει προσπαθήσει να στοχεύσει αυτά τα δύο πρόσωπα της κρίσης για να μπορέσει να εφαρμόσει πακέτα και ανακοινώσεις αρχέ, ε, τέλη Μαΐου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα αφορούν τη διάσωση ζωών και την μετακατάσταση 160.000 ανθρώπων από την Ιταλία και την Ελλάδα. Αυτά τα μέτρα εγκρίθηκαν άμεσα. Αρχές Οκτωβρίου έγινε μια συνάντηση εδώ στην Επιτροπή σας και σας έχουμε ενημερώσει από την DigiHome Home για την ανακοίνωση της 23ης Σεπτεμβρίου και συζητήσαμε και αυτές τις πρώτες δράσεις προτεραιότητας ε, τότε. Σήμερα λοιπόν έρχομαι να σας μιλήσω για την ανακοίνωση της 14ης Οκτωβρίου που παρουσιάζει ουσιαστικά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή αυτών των δράσεων προτεραιότητας. Όσον αφορά στα επιχειρησιακά μέτρα, τα πιο σημαντικά ε, στοιχεία είναι τα hot spots και το ε, σχέδιο μεταγκατάστασης έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά τα hot spots και την εφαρμογή των σχεδίων αυτών, των δύο σχεδίων, έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κοινή διαχείριση της κρίσης. Ε, το hot spot στη Λαμπεντούζα τώρα είναι πλήρως λειτουργικό και άλλα εγκαθίστανται πλέον στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα στη Λέσβο που σύντομα θα είναι λειτουργικό και έχουμε στοιχείο Σάμο, Κό και Λέρο άλλα τέσσερα και ελπίζουμε ότι αυτά θα λειτουργούν πλήρως μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται 105 άτομα μετεγκαταστάθηκαν από την Ιταλία και 30 από την Ελλάδα. Ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως πραγματικά πρέπει να επιταχυνθεί τώρα η διαδικασία. Αυτή η πρώτη εμπειρία ε, στην ουσία μας δίνει το σήμα για να μπούμε στην πρώτη φάση εφαρμογής. Ε. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για τις ε, προκλήσεις βάσει αυτών των πρώτων εμπειριών, γιατί ε, μιλάμε και για ε, αδυναμίες ε, πια. Έχουμε ανακαλύψει αδυναμίες σε αυτή τη φάση που σχετίζονται με το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή είναι απλώς στις απαρχές της. Πρέπει να μάθουμε πράγματα από αυτό, να ταυτοποιήσουμε τις προκλήσεις και να δουλέψουμε ώστε να τις αντιμετωπίσουμε με μεγάλη αφοσίωση. Ποιες είναι λοιπόν οι προκλήσεις. Καταρχάς η καταγραφή στην ανατολική πλευρά στον, ε, είναι πολύ χαμηλή ε, ε, γιατί το ΕΑΣΟ στην ουσία δεν έχει καλή, καλές επιδόσεις. 43% είναι η αντιμετώπιση των πρώτων αιτημάτων. Επίσης δεν υπάρχει και μεγάλη ανταπόκριση ως προς τα αιτήματα ασύλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε εσείς και εμείς να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Επίσης, ε, το, η πλήρης εφαρμογή των hotspot ε, στο ε, επόμενο, στο προσεχές μέλλον, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μπουν σε εφαρμογή οι μηχανισμοί ώστε η προθεσμία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενεργό δράση επιτόπου να μας βοηθήσει και να μας επιτρέψει αυτά τα hot να λειτουργούν μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου. όπως μας είπε το Συμβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς εσάς. Όμως ταυτόχρονα θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα από αυτή τη βραχυπροθεσμία αντίδραση και γι' αυτό ε, προτείναμε ένα μηχανισμό μετακατάστασης ε, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει διαρθρωτικά το θέμα της κρίσης, το θέμα του ασύλου. Αυτό το περιμένουμε να συζητηθεί. Το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη σε αυτό το θέμα και δεν χρειάζεται καν να σας ενθαρρύνω να ξεκινήσετε τη συζητήση για αυτό το θέμα το συντομότερο. Τώρα για άλλους τρόπους υποστήριξη των κρατών μελών γιατί η ανακοίνωση του Οκτωβρίου στην ουσία ακολουθεί τη δομή του Σεπτεμβρίου Και να, σε να σας ενημερώσω λίγο για τους τρόπους υποστήριξης των κρατών μελών που εμπλέκονται να σας ε, πω ότι όσον αφορά την παρουσία μας ε, στη θάλασσα αυξάνονται οι πόροι και τα κεφάλαια για τις ε, επιχειρήσεις της Frontex, Ποσειδών κτλ. Και τα κράτη-μέλη τώρα ε, πρέπει να δώσουν και αυτά επιπλέον πόρους ε, για αυτές ε, τις, τις επιχειρήσεις. Τώρα για την επιχείρηση γιονάτε περάσαμε από την πρώτη φάση αυτής της επιχείρησης που έχει να κάνει με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συλλογή δεδομένων. Στη δεύτερη φάση, αυτή η δεύτερη φάση έχει να κάνει με την με την ανοιχτή θάλασσα προσπαθούμε να πιάσουμε εκεί τους ε, λαθρέμπορους και να τους πάμε στη δικαιοσύνη. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της πολιτικής ασύλου και της επιχειρήσεις ε, της ε, ε, Frontex ε, είναι οι κοινέ επιχειρήσεις που έγιναν το 2015. Η Ιταλία συμμετείχε σε 10, η Ελλάδα σε 4 και οι βασικοί προορισμοί ήταν η Νιγηρία στο τέλος του έτους ε, θα έχουμε την αναθεωρημένη νομική βάση η οποία θα είναι εκεί για να βοηθήσει και τη διαχείριση των ε, συνόρων και την επιστροφή των άτυπων μεταναστών. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 και το σχετικό πρόγραμμα εργασίας. Και τώρα θα ήθελα να σας ε, αναφέρω κάποια ενημερωτικά όσον αφορά την συνεργασία με τρίτες χώρες. Και εδώ που γνωρίζετε από αρχάς Οκτωβρίου είχαμε αυτή τη συνάντηση ψηλού επίπεδου για Ανατολική Μεσόδιο και Βαλκάνια για να συζητήσουμε τι πρακτικά μέτρα μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τις χώρες εταίρων. Και ήταν πολύ σημαντική εκείνη η συνάντηση λόγω της ε, συμμετοχής αυτών των χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης ε, ε, σημαντικό ότι ήρθε η Τουρκία, η Ορδανία και ο Λίβανος και επίσης είχαμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που συζητήθηκαν και από αυτά που ανακοινώθηκαν που έχουν σημασία για την επιχειρησιακή υποστήριξη σε σχέση με Ορδανία Τουρκία και Λίβανο για τη διαχείριση της κατάστασης και του, των προσφύγων στις χώρες αυτές. Επίσης τέλος Οκτωβρίου έγινε συνάντηση κορυφής πάλι για τα δυτικά Κάνια όσον αφορά το ότι μετακινήθηκε η κρίση προς την Ανατολική Μεσόγειο και κατέληξε αυτή η συνάντηση ε, σε ένα πρόγραμμα 17 σημείων. Και αυτό είχε να κάνει με ψηφιακές ενέργειες οι οποίες ε, ανελήφθησαν ευθύς αμέσως. Uh, uh, uh, έχουμε τώρα σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα από αυτές τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις. Ότι δηλαδή έχουμε κάποιες τηλεδιασκέψεις σε όλες τις ε, χώρες με τα σημεία επαφής, αυτό γίνεται κάθε εβδομάδα και παρουσιάζουμε παρακολούθηση για τις ροές και αυτό ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Επίσης, ένα από τα ε, συγκεκριμένα σημεία αυτή της ε, ανακοίνωση αφορούσε το ότι θα αναπτυχθούν 400 αστυνομικοί στην ε, Σλοβενία. Και αυτό επίσης τώρα έχει υλοποιηθεί και επίσης τώρα έχουμε υλοποιήσει την καταγραφή των πόρων που έχουμε και την υποστήριξη από διάφορα χρηματοπιστωτικά εθελήματα διεθνή. Refer to Uh, point which Το um, uh, επόμενο σημείο αφορά αυτή την δήλωση ανακοίνωση όσον αφορά την εντατικοποίηση για τη συνεργασία με Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Αφγανιστάν και αυτά συμφωνήθηκαν. Και όσον αφορά τους επαναπατρισμούς. Επίσης, ε, έχουμε έκτακτη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών, η οποία έγινε και συζητήθηκαν όσα έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες. Συμφωνήθηκε επίσης να επιταχύνουν την υλοποίηση του γράμματος για τα hot spot και την επανεγκατάσταση. Και εν προκειμένου, τα κρατημέλη είπαν ότι θα κρατητήρισουν τις δεσμεύσεις τους ε, σχέση σχέση με την Frontex. Οπότε τα χθεσινά συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά από πλευρά του ότι έγινε μια καταγραφή της κατάστασης και επίσης έχουμε και κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία ενημερωτικής στρατηγικής, πως δηλαδή αυτή η στρατηγική θα πρέπει να αναβαθμιστεί για τους ετούντες άσου, τους πρόσφυγες, τους διακίνητες και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται ανάντι. Και να έχουμε επίση ενημέρωση των μεταναστών για τι υποχρεώσει τους και δικαιώματά τους και κυρίως για την υποχρέωση της καταγραφή τους στην πρώτη χώρα άφηξη. Και όπως είπαμε υπάρχει ε, προσοχή σε αυτό το τομέα, αλλά τώρα θα ενταθεί αυτή η πολιτική. Είπαμε να αναβαθμίσουμε την συνεργασία με την Τουρκία και θα πάει αυτή τη βδομάδα ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας εκεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κάποια συνάντηση για να δούμε πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Επίσης ε, δύο λόγια όσον αφορά το ζήτημα της χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Χωρίς να επισέλθω στις λεπτομέρειες, να σας πω ότι συζητηθήκε Θέλουμε να υπάρχει μια φυσιολογική δομή χρηματοδότησης. Με αυτό το ταμείο. Οπότε να υπάρχει συνεργασία και με τα εθνικά προγράμματα. Και επίσης να υπάρχει ενεργοποίηση της ε, βοήθειας σε κατεπήγοντα. και να εξεταστούν τα αιτήματα όπως έχουν αυτά υποβληθεί από τα κρατη Ελλάδα, Φινλανδία, Ουγγαρία είναι τα τελευταία αιτήματα που έχουν υποβληθεί. Οπότε και τα αιτήματα αυτά αξιολογούνται. Αφορούν περίπου 39 εκατομμύρια. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι που προβλέπονται για το όργανο το προενταξιακό για τις υποψήφιες χώρες. Αναφέρομαι σε Σερβία και Φιρόμ. Μιλούμε για κάποια ειδικά μέτρα 10 εκατομμυρίων. Αυτά έχουν προγραμματιστεί για διοικητικές, λειτουργικές ανάγκες αυτών των χωρών και για μη κυβερνητικού ε, οργανισμούς που δρούν εκεί. Επίσης έτσι προσπαθούμε να δούμε τι άλλα εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάποιες κατεπίγουσες καταστάσεις. Είπαμε για την πολιτική προστασία. Είναι κάτι που προέρχεται από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Πολιτικής και συνεχίζεται. Ε, το να βοηθήσουμε κάποιες χώρες που έχουν ανάγκη όπως Σερβία, Σλοβενία, Ουγγαρία και κάποιες αυτές τις χώρες καλύπτουν αυτό το μηχανισμό. Τώρα, πέραν της οικονομικής υποστήριξης και των οικονομικών εργαλείων που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση, έχουμε επίσης και κάποια καταπιστεύματα προβλέπεται ένα καταπίστευμα για την κρίση στην ε, Συρία και υπάρχει ένα άλλο για την Αφρική. Κατόπιν της συνάντησης κορυφής της Βαλέτας. Θα αρχίσουν αυτά να τρέχουν αυτή την εβδομάδα. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα εργαλεία, που είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλέπονται συγκεκριμένα κονδύλια, αλλά επίσης είναι σημαντικά γιατί είναι ανοιχτά στην ε, συμμετοχή και συμβολή των κρατών μελών. Οπότε και έτσι υπάρχει η δυνατότητα να αυξηθεί η πρικοδότηση. Τώρα, όσον αφορά την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου, ήδη τα είπαμε σήμερα το πρωί. Και στην ανακοίνωση μου βρείτε ένα παράρτημα το οποίο παραπέμπει σε κάποιες ε, υποθέσεις που αφορούν επαναπατρισμό και άσυλο. Και σας διαβεβαιώ και ως ε, φύλακα των συνδικών αλλά και ως Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών χρησιμοποιούμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και έτσι χρησιμοποιούμε τις νομοδιότητές μας και τις αξιοποιούμε. Επίσης βλέπουμε τι γίνεται με κάποιες παραβιάσεις του κοινωτικού δικαίου, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και τα βοηθάμε. Σε όσο γίνεται πρώιμη φάση για αυτές τις παραβιάσεις. Δηλαδή είμαστε σε συνεχή υπάρχουν τα κράτη-μέλη και ζητούμε πάντοτε συγκεκριμένες ε, ε, πληροφορίες, έχουμε δηλαδή ένα συνεχή διάλογο μαζί τους και όταν τα πράγματα γίνονται όπως πρέπει συνεχίζουμε δυνάμει των όσων προβλέπουν οι συνθήκες με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όσον αφορά την ενημέρωση και τα βασικά σημεία τα οποία περιέχονται στην ανακοίνωση τη Επιτροπής του Οκτωβρίου κατόπιν της προηγούμενη, αυτά ήθελα να σα πω. So I would like to thank you very much for Uh, your close involvement and, and cooperation. Uh, Επομένως βλέπουμε για στενή συνεργασία, ε, ενεργή εμπλοκή σας σε όλα αυτά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ε, κάνουμε βήματα πρόοδου σε σχέση με τα νομοθετικά θέματα τα οποία εκκρεμούν και ό,τι άλλο μας υποβληθεί. Οπότε και βέβαια είμαστε και στην ε, διάθεσή σας να ακούσουμε τι παρατηρήσεις έχετε που είναι σημαντικές για μας γιατί ξέρουμε ότι έχετε πολλές επαφές και πηγές επιτόπου και ότι έχετε επισκεφθεί ε, τις, τις επίμαχες περιοχές οπότε υπάρχουν πληροφορίες που μπορείτε να μας δώσετε για να δούμε τι συμβαίνει πάντως εγώ στέας διαβεβαιώνω ότι όλοι οι συνάδελφοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση Ελπίζουμε να υπάρξει μια λύση το συντομότερο δυνατόν, αλλά δεν πρόκειται για μια αντεπροσβευτική κλασική κρίση. Θα πάρει λίγο παραπάνω αυτή η κρίση. Οπότε πάντως ε, αυτή, αυτή είναι η γενική άποψη που έχουμε και το θεματολόγιο μας. Δεν είναι μόνο θέμα του κατεπήγοντος νομίζω ότι το κοινό μας έργο μέσα από αυτή την εμπειρία πρόκειται ε, να μας κάνει να βγούμε κερδισμένοι και ούτω ώστε αργότερα θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη μετανάστευση καλύτερα. Άρα είναι κάτι που πάει πιο πέρα από την βραχυπρόθεσμη προοπτική. Είναι κάτι μακρόπνο. Επομένως καλή τύχη, σε όλους μας καλή επιτυχία. Και με ενδιαφέρουν οι παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε ως προς την εφαρμογή των μέτρων της Κομισιόν. Αρχίζουμε τώρα με τον κύριο Γκαρσία Ντεμέρα. Muchas Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την ενημέρωση της κυρίας Σιγκάν και Έχω πολλές ερωτήσει να υποβάλω, αλλά από όλε αυτές μία τελικά θα σα πω. Και δεν ξέρω αν αυτό γίνεται επίτηδες ή επειδή τα μαντάτα δεν είναι και τόσο ορόδινα. Και άκουσα όλα αυτά που μας είπε. Γιατί άκουσα για επανεγκατάσταση, αλλά για μετεγκατάσταση. Οπότε Μπάς και μπορείτε να μας ενημερώσετε για την κατάσταση. Για το τι γίνεται με αυτή την μετακατάσταση. Και τι δυναμική υπάρχει. Γιατί έχουμε 20.000 επανεγκαταστάσεις και πολύ λιγότερες μετακαταστάσεις. Και αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία λίγο πολύ είναι στον χώρο του φανταστικού. Οπότε για πέστε μας κάτι συγκεκριμένο. Εγώ αυτό χρειάζομαι. Αλλά και νομίζω θέλουμε όλοι να μάθουμε τι γίνεται όσον αφορά την μετακατάσταση. Ευχαριστούμε κύριε Ντεμέρα. Σιλβί Γκυγιόμ των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου για αυτά που μας είπατε για το μεταναστευτικό. Έχουμε την εντύπωση ότι ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να συζητιούνται. Τώρα όμως πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά συγκεκριμένα. Γι' αυτό είναι καλό που μας δώσατε μερικές αποσαφηνήσεις γιατί επίσης έχουμε την εντύπωση ότι αρχίζει κάποια δράνεια. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να προχωρήσουμε και ο πρώτος αντιπρόεδρος της ε, Κομισιόν μας είπε το ιστορικό Winter is coming. Επομένως πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Τέσσερα πρόσθετα αιτήματα πληροφόρησης έχω. Πρώτον, τα hot spots που για μένα είναι, παραμένουν ανησυχητικά. Μας δώσατε μερικές πληροφορίες αλλά θα ήθελα να ξέρουμε συγκεκριμένα πώς λειτουργούν αυτά. πώς γίνονται οι καταγραφές ε, κλπ. στα hot spot. Επίσης είδα ένα ρεπορτάζ της προάλλες στη Γαλλία για το σύστημα της εγγραφής των προσφύγων και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ένα διπλό σύστημα, το επίσημο και το ανεπίσημο. Δεν κατάλαβα αν αυτό οφείλεται, αυτό το κάνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή οι ελληνικές αρχές, αλλά ότι είναι λέει λίγο πιο ταχύ και λίγο πιο γενικό. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Έπειτα. Μπορείτε να μας πείτε τίποτα για τις μετεγκαταστάσεις, για τις ε, επιστροφές και γι' αυτό μερικές λεπταμέρειες. Και τέλος, αν και είναι μόνο το τρίτο σημείο, τα πρόσθετα μέτρα για το δικαίωμα ασύλου τι συνέχεια δόθηκε. Αν έχετε καμιά παρατέρω λεπτομέρεια και τελευταίο το τέταρτο πάλι τελευταίο, είπατε ότι η δυσκολία λέει είναι ότι μερικοί που ετούνται άσυλο δεν έχουν δικαίωμα σε αυτό γιατί δεν προέρχονται από τρίτες χώρες που καλύπτονται από συμβάσεις. Αυτό κατάλαβα. Η κυρία Βίξτρομ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είναι πάντοτε ενδιαφέρον να συζητάμε αυτά τα θέματα αν και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν η αξιοπιστία της Ένωσης που αμφισβητείται συνεχώς. Οι αριθμοί ανθρώπων που μεταφέρονται από τις μετεγκαταστάσεις είναι χελιοδός χαμηλή προς το παρόν. Θα ήθελα να γνωρίσω γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό σε τι οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις. Γιατί πάλι αποτυγχάνουν τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν υπογράψει. Και τι σχεδιάζει να κάνει η Κομισιόν ώστε οι μετεγκαταστάσεις να εφαρμόζονται σωστά στη Σουηδία. Όπως ξέρετε δεχόμαστε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Μέχρι τώρα 190.000 περίπου που είναι παραπάνω από 160.000 υψηλότερος αριθμός από το μερίδιο που μας αναλογούσε. Άρα δεν πρόκειται για λογικό επιμερισμό ευθυνών και θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν τι θα κάνει τώρα ως προς το αίτημα της Σουηδικής Κυβέρνησης για συμμετοχή στις μετεγκαταστάσεις ώστε να βοηθηθεί η Σουηδία να μεταφέρει πρόσφυγες και από τη Σουηδία σε άλλες χώρες. Αυτό ζητάνε οι πολίτες στη χώρα μου. Και θέλω πραγματικά να μου πείτε, να μου απαντήσετε, τι θα κάνει η Κομισιόν γι' αυτό. Τι. Κυρία Φεράρα. Πού είναι, δεν είναι εδώ, Ευχαριστώ πρόεδρε, ναι. Ε, βέβαια και ακόμα είμαστε μακράν το να πετύχουμε αυτές τις ε, πρωτοβουλίες όλα αυτά τα οποία είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε φρένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, οπότε δεν πάμε προ τα εκεί που θέλαμε να έχουμε κατευθυνθεί. Οπότε και ακόμα περιμένουμε τις προτάσεις με την ε, τροποποίηση της συνθήκης του ε, Δουβλίνο. Αυτό χρειάζεται να γίνει γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε και έτσι να μπορούμε σε σχέση με την πρώτη χώρα υποδοχής να ε, έχουμε τις ευθύνες όλες τις ρυθμίσεις ειδικά με την υποδοχή και ακόμα επομένως έχουμε πολλές ε, επιφυλάξεις όσον αφορά το πώς θα ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση και τι ευθύνες θα αναλάβουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν πολύ σκεπτικισμό ακόμα σε σχέση με αυτό και άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και έτσι δεν επιδεικνύουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την διαχείριση των ροών, την αλληλεγγύη που θα έπρεπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την κρίση του μεταναστευτικού και μόνο ένα συμπέρασμα μπορώ να βγάλω. Δεν υπάρχει στην ουσία απάντηση. Έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες σύνοδοι κορυφή, όμως ε, ένα χάος δημιουργήσαμε περισσότερους ετούντες άσυλο. Και αν δούμε τα χθεσινά νούμερα θα καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα που αυξάνεται και δεν διαφαίνεται το τέλος. Αυτή η κρίση για άλλη μια φορά ξε... μας ε, δείχνει ότι οι εκλεγμένοι γραφειοκράτες της Βρυξέλλες δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι έχει χρεοκοπήσει το Σέγγεν. Πρέπει να κλείσουν τα σύνορα. Η μετανάστευση είναι ένα εθνικό θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κρατήσει τα χέρια της μακριά από αυτό. Έχω ένα ερώτημα. Ξέρω ότι ε, υπάρχει μια αντιπροσωπεία που θα πάει στην Τουρκία για συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να μας πείτε είτε στην ουσία τι ακριβώς θα διαπραγματευτούν και πότε πρέπει να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που φτάνουν στην Ελλάδα και την Ιταλία και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ε, για τη μετακατάσταση. Ε, πού πηγαίνουν, πηγαίνουν σε τρίτες χώρες, πηγαίνουν στην χώρα προέλευσής τους. Ευχαριστώ κυρία Σπινιέλη. Πριν μιλήσουμε για τα hotspot και τα προβλήματα τα σχετικά, να δούμε ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή κατάσταση και θέλω να επισύρω την ε, προσοχή της Επιτροπής όσον αφορά την αρρωγή προς την Ελλάδα. Η Επιτροπή λέει ότι θέλει να τηρήσει την δέσμευση σε σχέση με την αρρωγή προς ε, κάποια χώρα η οποία βρίσκεται υπό πίεση των μεταναστευτικών ροών που όλοι τις γνωρίζουμε. Πάντως, εδώ συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχει αναφερθεί η Ευρωπαϊκή Εντροπή σε αυτές, ούτως ώστε να υπάρξει χρήση ε, των δυνατών των σχετικών κονδυλίων. Μα για ποιους όρους και προϋποθέσεις μιλώ. Οι ελληνικές αρχές έχουν κλείθει να μπορέσουν να παράχουν πρώτα-πρώτα κάποιες υπηρεσίες. Καθαριότητα, τρόφιμα, κέντρα υποδοχής κλπ. Οπότε κατόπιν προβλέπεται να λάβουν τα χρήματα. Όμως μετά από τόσα χρόνια λιτότητα στην Ελλάδα αυτή η ρυθμίση του πρόσωπου Ευρωπαϊκής δείχνει μια τέλεια άγνοια της κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι σε θέση του να προκαταβάλει αυτά τα χρήματα. Βεβαίως και υπάρχουν λύσεις, λύσεις ρεαλιστικές. Δηλαδή το να μπορέσει να έχει αυτά τα χρήματα η Ελλάδα σε κάποιον λογαριασμό για να γίνει άμεση χρήση αυτών των χρημάτων άπαξ και κριθεί ότι συντρέχει λόγος κάποιας παροχής υπηρεσίας και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να μπορέσει να υπολογίσει τα σχετικά έξοδα υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται όμως για ένα ζήτημα επίγον κυρία, κυρία Σίγκαν. Οπότε θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση ακριβή, μια που πρόκειται για θέμα κατεπίγον. Τώρα, για τα σημεία υποδοχή, τα hot spots. Όχι, δεν έχω χρόνο. Ναι, ναι, να μου δώσετε το χρόνο, ωραία. Στην Ιταλία έχουμε τα hot spots και εκεί λέτε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εγγυηθούμε κάποιους ειδικούς από την ΕΑΣΟ και από την, ε, και από την ε, Frontex ούτω ώστε να μπορέσουμε αυτά τα κέντρα να τα έχουμε για να καλύψουμε κάποιες μεγάλες ε, περιόδους και ταυτόχρονα να είναι έτοιμα αυτά τα κέντρα όσο γίνεται πιο σύντομα. Οπότε, να ρωτήσω την Επίτροπο της Επιτροπής, αφού λέμε ότι θα επιστρατεύσουν αυτά τα κέντρα για μακρά περίοδο, Οπότε θα πρέπει επομένως τα σημεία υποδοχές να διέπονται από το άρθρο 78 της συνθήκης για τα θέματα τα κατεπήγοντα. Και άρα θα πρέπει να υπάρξει και κάποια ρύθμιση πάγιο χαρακτήρα για ζητήματα κατεπήγοντα. Ε, οπότε θα πρέπει επομένως έτσι να έχουμε αυτά τα κέντρα τα οποία να λειτουργούν επαγίως χωρίς να χάνουν τον κατεπήγοντα χαρακτήρα αντιμετώπισης. Τι πάει να πει αυτό. Το ότι θα έχουν αυτό το χαρακτήρα και θα πρέπει να ληφθεί κάποια απόφαση αλλά θα ληφθεί μονόπλευρα. Δεν θα συμμετέχει σε συναπόφαση το Κοινοβουλίο. Θα λάβει την απόφαση μόνη της, τελείως μόνη της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ βάζω τελείω γιατί σας είπα πολλά. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να σέβεστε όλοι τον χρόνο ομιλία στο πολύ δύο λεπτά. Τώρα η κυρία Χιμένες, αν δεν απατώμε. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω, πολλά ήδη ρωτήθηκαν, αλλά θέλαμε κάποια ενημέρωση παραπάνω σχετικά αφορά αυτό το μητρό, το μητρό καταγραφής των ε, προσφύγων. Πώς είναι, τι γίνεται, να λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα, ε, από την άλλη μεριά δεν τα δίνουν, ε, δεν συνεργάζονται γιατί φοβούνται ότι τους διώξουν από τη χώρα υποδοχή Ενώ βέβαια υπάρχει το δικαίωμα ετήσεως ασύλου στην χώρα υποδοχής. Θέλουμε επομένω να υπάρχει στο κέντρο αποδοχή να προβλέπει κάποια διάρκεια 8 μηνών ή παραπάνω και έτσι να λυθεί το πρόβλημα ακριβώ αυτό που είπε η κυρία Φεράρα και έτσι η Ελλάδα και η Ιταλία να ανακουφιστούν γιατί έχουν ε, αναλάβει όλο αυτό το βάρο μέσω των hot spots. Να δούμε πώ μέσω τη αλληλεγγύης θα βοηθηθούν αυτέ οι ε, χώρες. Μα πώς, πώς θα γεμίσουμε τις χώρες αυτές με hot spots αφού δεν υπάρχει οικονομική υποστήριξη. Πώς θα το αναλάβουν αυτό αυτές οι χώρες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αυθεντικές μετεγκαταστάσεις γίνονται πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό και πάρα πολύ με προβληματίζει το τι θα πει για εκείνη γνώμη για αυτά τα κέντρα κράτησης, εγκατάστασης, τέλος πάντων τα κλειστά. Έρχεται τώρα ο χειμώνας και όλοι αυτοί οι πρόσφυγες τι θα κάνουν μόλις φτάσει η κακοκαιρία γιατί θα γεμίσει ο κόσμος από αυτές τις φοβερές εικόνες της τηλεόρασης. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα θέματα. Πρώτον, Διάβασα στην εφημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Κομισιόν λέει έχει λάβει 3 εκατομμύρια πρόσθετων ετοιμάτων ασύλου από το 7 σε σύγκριση με το 7. Είναι ισχύει αυτή η πληροφόρηση και αν ναι τι θα κάνετε. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, για τα hot spots οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι ότι πολλοί πρόσφυγες αρνούνται να εγγραφούν στα hot spots. Τι θα τους κάνουμε αυτούς, τι θα απογίνουν, τι πολιτική θα εφαρμόσουμε για αυτούς. Είπατε επίσης, δεν κατάλαβα ποιον στοχεύατε όμως, ότι μερικοί λέει δεν προέρχονται από χώρες που προβλέπονται, τι θα πει αυτό που προβλέπονται. Τρίτον, για τα ταμεία μιλήσαμε πολύ, αλλά δεν παίρνουν τίποτε τα κράτη-μέλη. Πληρώνει η Ένωση ό,τι είχε προβλεφθεί, αλλά ποια είναι η στρατηγική της Κομισιόν για να οθήσει τα κράτη-μέλη, δεν ε, πληρώνουν τα κράτη-μέλη, να πληρώσουν. αφού γίνεται λόγος για κινητοποίηση και άλλων ποσών ακόμη και ιδιωτικών. Τέταρτο, πότε ακριβώς προβλέπετε να υποβάλλετε ένα νέο νομικό υπόβαθρο για το Frontex. Γιατί λέτε ότι θέλει να επεκταθεί η εντολή του. Φαντάζομαι για να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στα hot spots και για τις μετεγκαταστάσεις ή τις επιστροφές. Πότε ακριβώς το προβλέπετε αυτό να αλλάξει το νομικό υπόβαθρο και να το υποβάλλετε στην Επιτροπή μας. Αυτά. Ευχαριστούμε κύριε Ντεπρέ. Η κυρία Κέλλερ τώρα, η ΣΚΑ. Ξέρετε ότι ήταν και η συγκήτρια. Απαντήσω σε μερικά από αυτά που ρώτησε ο κύριος Ντεπρέ Μίλησε για εκείνους που δεν θέλουν να εγγραφούν. Αντίθετα, εγώ βλέπω ότι υπάρχουν ουρές για να εγγραφούν και δεν υπάρχει χώρος. Όλοι θέλουν να εγγραφούν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν πάντοτε, εκτός αν δεν κατάλαβα καλά. Πώς, πώς. Προσπαθούν να εγγραφούν παντού. πάντε πηγαίνετε και κοιτάξτε προσπαθούν να εγγραφούν στο hot spot αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις και δεν μπορούν να εγγραφούν όλοι. Μήπως δεν κατάλαβα καλά, μήπως έγινε λάθος μετάφραση. Τώρα, γιατί δεν μετεγκαθίστανται, αυτό εξαρτάται γιατί μερικές χώρες δεν εφαρμόζουν τις υποσχέσεις τους. Ας πούμε η Γερμανία μπορεί να προσφέρει 10 θέσεις ενώ μπορεί να υπάρχει 12 μελής οικογένεια. Υπάρχει όμως και άλλο προτεραιότητες των προσφύγων δεν λαμβάνονται υπόψη. Καθυστερούν τα κράτη-μέλη μέχρι να αποφασίσουν ποιος θα πάει πού. Καθυστερήσεις μέχρι και δύο μηνών. Τους λένε ότι μπορεί να εγκατασταθούν σε κάποια χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί επιχόντως. Ερωτώ δε την Κομισιόν τι προτείνεται για την νόμιμη και ασφαλή είσοδο των προσφύγων, γιατί ξέρετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, η θάνατη στη θάλασσα κτλ. Επίσης, μπορεί να θυμάστε ότι είχαμε δώσει περισσότερα χρήματα στο Frontex για να μπορεί να σώζει περισσότερους στη θάλασσα. Τους δώσαμε τα λεφτά χρησιμοποιούνται για περισσότερα πλοία αλλά όχι για περισσότερες διασώσεις. Γιατί το Frontex επιτηρεί απλώς και ζητάει από την τουρκική ας πούμε αστυνομία να επιστρέψει τους ε, πρόσφυγες. Αυτό δεν είναι σωστό. Το Frontex δεν πρέπει να σώζει όποτε τύχει, αλλά να είναι η κύρια του αποστολή. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλερμα. Τώρα η κυρία Γουίνμπακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά με ανησυχεί το θέμα της χώρες μου. Η κυρία Βίξτρομ είπε ότι 190.000 έρχονται προς την Σουηδία και ε, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός ε, της ε, Σουηδίας ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει πίσω τους 50.000. Πραγματικά μπορεί να η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας λέει τι θα κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Γιατί ενδεχομένως τώρα να έχουμε ένα κόμμα το οποίο θέλει να εισαγεί ελέγχους, όμως ε, ε, πραγματικά η όλη η ιστορία στη Σουηδία είναι τελείως διαφορετική. Ε, πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι η Σουηδία έπρεπε να πάρει κάποια άτομα και τελικά πήρε μόνο πολύ λίγα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έρθουν στη χώρα μας και περνάνε από άλλες χώρες ε, και οι, ίδιοι ε, ενδεχομένως αποφασίζουν ε, που θέλουν να πάνε. Αυτό το έχουμε σκεφτεί για τα ταμεία τώρα και στα ταμεία ρίχνουμε ένα σωρό χρήματα. Έχουν τα κράτη-μέλη χρήματα να βάλουν σε αυτά τα ταμεία. Αν πρέπει να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη μαζική μετανάστευση τα κράτη-μέλη πραγματικά θα γονατίσουν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει κάπως να ξανασκεφτούμε τα πράγματα. Χρειαζόμαστε φυσικά να δώσουμε βοήθεια σε κάποιους, σε κάποιους να υποστηρίξουμε, ε, αλλά πραγματικά τι θα κάνουμε για να λύξουμε αυτή την κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να βρούμε. Ε, ευχαριστώ, θα ήθελα ε, να διαμαρτυρηθώ γιατί πήρα το λόγο μετά από τη Σουηδή συνάδελφο πραγματικά που εκπροσωπεί το μικρό, τη μικρότερη ομάδα και την ακροδεξιά της Σουηδίας ενώ εγώ ανήκω στην πιο μεγάλη πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να χαιρετήσω την δέσμευση της Κομισιόν ε, για το θέμα της ε, μετανάστευσης επίσης για την ε, στεναρή απάντηση του Γιούνκερ και την προσπάθεια που κάνει, παρόλο που υπάρχει έλλειψη ε, ε, εφαρμογής των ε, μέτρων που λαμβάνονται, 160.000 είναι οι άνθρωποι που θα μετεκατασταθούν, μεταξύ αυτών ελάχιστοι από την Ιταλία στη Σουηδία. Δεν ξέρω πότε μπήκε η Σουηδία στον χάρτη. Πραγματικά η κατάσταση είναι έκτακτης ανάγκης στο Γκέτεμπουργκ και υπάρχουν άνθρωποι που σε σκηνές καλωσορίζουν κόσμο. Στο Μάλμο επίσης με τα τρένα φτάνουν άνθρωποι και υπάρχουν ε, πραγματικά συνόδευτοι ανήλικοι που χρειάζονται περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Και το σύστημα της Σουηδίας που είναι ένα από τα καλύτερα δεν μπορεί να ε, ανταποκριθεί πλέον φυσικά. Ε, δεν ζητά βοήθεια η κυβέρνηση, όμως ε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί όλα τα ε, επιπλέον μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν να κάνουν με τις χώρες της πρώτης υποδοχής που έχουν ε, σύνορα με τρίτες χώρες και με τις χώρες διαμετακόμισης και όχι με, με μας. Οι άνθρωποι λοιπόν που έρχονται δεν δακτυλοσκοπούνται η Σουηδία στην ουσία ε, έχει γίνει χώρα πρώτης υποδοχής και χώρα τελικής υποδοχής ε, παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από άλλα κράτη-μέλη και έχουμε μία δυσανάλογη πίεση στα ε, σύνορα και τις μακροπρόθεσμες φυσικά προκλήσεις σε επίπεδο αγοράς εργασίας, στέγασης και φυσικά εκπαίδευσης των παιδιών. Τα ζητήματα λοιπόν είναι πολλά και τα ερωτήματα πολλά προς την Κομισιόν. Θέλετε να βάλετε και την Σουηδία στο ε, σύστημα μετακανάστασης των 160.000. Ναι, ε, παρόλο που η Ουγγαρία δεν θέλει να συμμετάσχει, θα μετέχει η Σουηδία στα μετολικά συστήματα μετακατάστασης. Θα έχετε hot spots και για τη Σουηδία. Έχετε επιπλέον μέτρα που θέλετε να θεσπίσετε για να αντιμετωπίσετε το θέμα των ασυνόδευτων μεταναστών που χρειάζονται επιπλέον πόρους. Έχω άλλη μία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, σχετικά με το ε, σχέδιο του καρότου, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι. Ο κύριος Γιούγκερ είπε στην Ολομέλεια ότι οι χώρες της Ευρωζώνης που θα δείξουν ότι καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες στο θέμα της μετανάστευσης θα έχουν τη δυνατότητα ευέλικτης ε, ερμηνείας του ε, Συμφώνου σταθερότητα. Τι γίνεται τώρα με τις χώρε που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Δεν είναι αυτό διάκριση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο τα μέλη της Ευρωζώνης δέχονται ε, εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις. Τι θα γίνει με τα μη ε, μέλη της Ευρωζώνης. Θα κάνει η Κομισιόν κάτι. Ε, για το θέμα των τον άσυλο, πώς θα αντιμετωπιστεί ε, το τεράστιο νούμερο τέτοιων ανθρώπων που ήδη γίνονται αποδεκτοί. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, μπορεί η Κομισιόν να μας πει αν θα δημοσιεύσει την κατανομή των οικονομικών, ανθρώπινων και άλλων διοικητικών πόρων που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές στη Συρία, στην Αφρική κτλ. Γιατί πρέπει πραγματικά να κατονομάσουμε και να το πιάσουμε τα κράτη-μέλη που εμπλέκονται. Ευχαριστώ. Έχετε μιλήσει δύο φορές, περισσότερο από τους υπόλοιπους, να σας πω. Ο κύριος Κοέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις δηλώσεις. Ε, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ με την ιδέα της κυρίας Καγενότη που λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη ανάγκη, αλλά δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε την πηγή του προβλήματος και τα μακροπρόθεσμα μέτρα υπογραμμίσω αυτό που είπε η Σεσίλια Βίξτρομ. Δεν καταλαβαίνω και το Κοινοβούλιο δεν καταλαβαίνει πώς μιλούν τόσο πολύ τα κράτη-μέλη για μεγαλύτερη διασφάλιση των συνόρων, αλλά δεν δίνουν αρκετούς ανθρώπινους πόρους ε, για να ε, καταγράφονται και να ε, ελέγχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στα σύνορα. Υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο αριθμό μεταναστών και οι αποφάσει δεν είναι στο των περιστάσεων. Γιατί διατηρούμε ε, όλους αυτούς τους συνοριακούς ελέγχους όταν μόνο 160.000 από τους 90 ε, από τους 900.000 ε, μετανάστες και πρόσφυγες θα μετεγκατασταθούν. Υπάρχουν τα θέματα της μετεγκατάστασης μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικά και άλλα θέματα αλληλεγγύης. Ας πούμε στη χώρα μου πολλά ΜΚΟ οργανώνουν δίκτυα υποδοχής αυτών των ανθρώπων και τώρα δεν φτάνουν οι πόροι, τα πάντα βρίσκονται στον αέρα. Υπάρχει αυτή η απογοήτευση και η ιδέα ότι η Ευρώπη δεν λειτουργεί και γι' αυτό ανησυχώ. Τώρα για τα hot spots. Όταν και αν πάνε αξιωματούχοι της ΕΑΖΟ στην Ιταλία και την Ελλάδα, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν πάνε, υπάρχει έλλειψη ε, στο διάστημα ε, μέχρι την 9η Νοεμβρίου, 4 με 9 Νοεμβρίου, 90.000 ε, άνθρωποι έφτασαν στην Ελλάδα. 6.000 την ημέρα δηλαδή μπορούν τα hot spot να καταγράψουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται και άλλα κέντρα υποδοχής. Επίσης, ένα πιλωτικό project για πιο γρήγορη ε, δήλωση ε, εισόδου ε, γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μπορεί να πετύχει. Η Σιλβί Γιόμ ήδη μίλησε για την επιστροφή στις χώρες προέλευσης. Κατάλαβα ότι η Κομισιόν θα καταθέσει μία πρόταση για διεύρυνση των επιχειρήσεων της Frontex σε αυτό το επίπεδο. Περιμένουμε την πρόταση. Όμως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συμφωνία για να μπορέσουμε να ε, στείλουμε πίσω στις τρίτες χώρες τους ανθρώπους αυτούς. Η Κομισιόν κάνει κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Αλάου από το ECR. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Την τελευταία δήλωση του Συμβουλίου μεταξύ άλλων λέει και αναφέρω πρέπει να εξηγηθεί ξεκάθαρα στους μετανάστες ότι πρέπει να δηλώσουν την είσοδό τους στο πρώτο κράτος μέλος ε, αφήξης και δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το κράτος μέλος που θα εξετάσει την αίτησή τους. Τώρα το ερώτημα είναι ενδιαφέρον. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη εάν και όταν τα οι μετανάστες δεν εγγραφούν στο πρώτο κράτος αφήξης. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει ένα κύμα μεταναστών σε όλη την Ευρώπη που πηγαίνουν προς τη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Για παράδειγμα, η Σουηδία θα πρέπει να αρνηθεί αιτήματα από ανθρώπους που έρχονται από τη Δανία ή η Φιλανδία από τους δεκάδες χιλιάδες που έρχονται από την Σουηδία. Αυτή τη στιγμή τα αιτήματα αυτά είναι υπό επεξεργασία και φαίνεται μάλλον γελίο να λέμε στους μετανάστες ότι υπάρχουν κανόνες όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Μπιόκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη. Έχουν ήδη υποθεί πολλά. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε και η κυρία Σπινέλη για την Ελλάδα οι πόροι δεν φτάνουν στη χώρα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και δεν αρκεί να λέει η Κομισιόν ότι να έχουμε αποφασίσει να δώσουμε τα χρήματα. Τα χρήματα δεν έχουν φτάσει εκεί. Ε, πώς θα αντιμετωπιστούν όλοι οι άνθρωποι που ε, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν από το κρύο. Για τη Frontex. Η κυρία Κέλλερ είπε ότι... Ε, ε, έχουν δοθεί επιπλέον μέσα ε, για να ε, μπορέσουν να διασωθούν άνθρωποι στη θάλασσα, αλλά αυτό δεν γίνεται και χρειάζεται τα ψαροκάικα στην Ελλάδα να σώζουν τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά σκάνδαλο που πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι στην Μεσόγειο. Για τα hot spot χρειαζόμαστε συγκεκριμένη αντιμετώπιση, ε, πρέπει να δούμε πώς ακριβώς ε, θα πρέπει να λειτουργήσουν και θα ήθελα πραγματικά να συζητήσουμε και το θέμα του προϋπολογισμού, των κονδυλίων. Ε, πραγματικά χρειάζεται μεγάλη διαφάνεια σχετικά με το πού πηγαίνουν τα χρήματα. Η Κομισιόν τελικά έχει καταλάβει ότι πηγαίνουν τόσα χρήματα σε κατασταλτικά μέτρα στους ελέγχους των συνόρων. στην εκπαίδευση των διαφόρων ε, δημοσίων υπαλλήλων ε, που ε, εργάζονται σε τρίτες χώρες στο θέμα της μετανάστευσης, όμως τελικά το πόσα χρήματα δίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις στο κάτω-κάτω της γραφής για τη μετανάστευση δεν είναι ξεκάθαρο. Εμείς είμαστε μια χώρα που είναι καλά οργανωμένη, υπάρχει ευημερία, υπάρχει αλληλεγγύη, έχουμε μεγάλο ε, αριθμό ε, προσφύγων, υπάρχουν κάποια κόμματα πολιτικά που θέλουν να το σταματήσουν αυτό, όμως ε, τα καταφέρνουμε. Χρειαζόμαστε παρόλα αυτά ένα συγκεκριμένο σχέδιο όσον αφορά στην απασχόληση, την στέγαση, την εκπαίδευση, να είναι μακροπρόθεσμο και να δίνει πρόσβαση στον κόσμο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν ε, όσον αφορά στη συνεργασία με τα διάφορα γραφεία και τους οργανισμούς ας πούμε του ΟΗΕ ε, πώς θα προχωρήσει. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και χρειάζεται να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο και Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, οπότε και εγώ θα περιοριστώ σε λίγες ερωτήσεις. Λίγες αλλά σημαντικές. Δεν ξέρω γιατί καλύπτουμε τώρα μόνο Ελλάδα και Ιταλία με αυτά τα μέτρα γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε πιο ευρύ αντιμετώπιση και να καλύψουμε και άλλες χώρες. Γιατί αυτό τα στοιχεία το μας δώσανε δεν είναι ενημερωμένα, δεν αντικατοπτρίζουν τη σημερινή κατάσταση. Σήμερα δε έχουμε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει στο Αφγανιστάν και έχουμε 70.000 Αφγανού οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα του τι τελευταίε τρει εβδομάδε. Όλοι αυτοί κατευθύνονται προ την Ελλάδα, ήρθαν στην Ευρώπη και τι θα γίνει με την Τουρκία, γιατί στο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα η κατάσταση αυτή είναι δεν υπάρχει τίποτα για Σουηδία, Ουγγαρία, Κροατία. Θα πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και μας πείτε πώς έχει η κατάσταση σε όλες αυτές τις άλλες χώρες. Κάποια άλλη ερώτηση τώρα όσον αφορά κάποιον μηχανισμό για την επανεκατάσταση των προσφύγων τι θα γίνει, θα υπάρξει τέτοιος μηχανισμός τελικά, γιατί το σημερινό σύστημα σαφώς δεν αποδίδει, δεν επαρκεί. Έχετε κάποιο πρόγραμμα. Τι είδους πρόγραμμα είναι αυτό. Τι θα κάνει η Επιτροπή ούτως ώστε να εξασφαλίσει ότι η Γερμανία και η Σουηδία θα αλλάξουν το σύστημα της κοινωνικής προνοίας τους για να αντιμετωπίσουν όλους αυτούς οι οποίοι ετούν άσυλο θα γίνει με την Τουρκία επίσης. Έχουμε 25.000 διακινητές οι οποίοι δρούν στην Τουρκία. Πότε θα αντιμετωπιστούν. Τι γίνεται με τις ασφαλείς χώρες, γιατί ορισμένα γερμανικά δεστηρία δεν αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως ασφαλή χώρα. Πότε θα δούμε ε, τον οριστικό κατάλογο των ασφαλών χωρών. Αφγανιστάν και Πακιστάν θεωρούνται ασφαλείς χώρες. Επίσης, τι γίνεται με το κοινό σύστημα για το άσυλο. Χαίρομαι που το αναφέρατε, αλλά έχω να σας πω το εξή. Ο λόγος που ο κόσμος αποφεύγει τα hot spots είναι το ότι γνωρίζουν πως έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν άσυλο σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και χρειάζεται συζήτηση πιο ενδελεχής για την πολιτική του ασύλου. Κυρία Ζολή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να μας πει η Κομισιόν δύο πράγματα. Τα τρία τελευταία χρόνια ασχολήθηκα πολύ με το Αφγανιστάν και έχω πάει επανειλημμένο στην Καμπούλ. Και θα ήθελα να μας, διαβεβαιώσουν, να μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα επιστραφούν Αφγανοί στο Αφγανιστάν με την πρόφαση των ασφαλών χωρών. Όταν φεύγουν τσάρτερ από τις βόρειες χώρες ή την Αγγλία φτάνουν στην Καμπούλ χωρίς καθόλου λεφτά. Οι περισσότεροι δεν προέρχονται από την Καμπούλ αλλά από το Χεράτ, το Τζαλαλαμπάντ και αλλού και δεν είναι ασφαλείς οι δεν μπορούν να φύγουν μετά από την Καμπούλ και μετά από τρεις-τέσσερις μέρες γίνονται λία εκμετάλλευσης από τους Ταλιμπάν. Κάναμε τον πόλεμο τόσα χρόνια στο Αφγανιστάν για να αφήσουμε τους ανθρώπους που έρχονται από εκεί και συνήθως νέους στα χέρια των Ταλιμπάν. Παράλογο. Έπειτα. Θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι δεν θα συστήσετε στο Συμβούλιο την επανάληψη των διαδικασιών του Δουβλίνου γιατί η Ελλάδα δεν έλαβε τα 2,5 δισεκατομμύρια βοήθειας που υποσχεθήκατε τον πρόσφατα. 150.000 το μήνα ανθρώπους δέχεται η Ελλάδα και θα ήταν παράλογο να επανεγκατασταθούν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες με το πρόσχημα της διαδικασίας του Δουβλίνου. Ευχαριστούμε. Λουρέκ. Λουρέκ. Ευχαριστώ. Έχω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα, λέω ο κύριος Γιούρεκ. Πρώτον, Γιατί είναι τόσο βραδία η πρόοδο στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της διακίνησης αυτών των μεταναστών. Υπάρχει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορά τα χωρικά έδατα της Λιβύης. Αλλά, όπως είπε κάποιος συνάδελφος τώρα καινούργιες διαδρομές ξανοίγονται μέσα από την Τουρκία μέσω της Μαύρης Θάλασσας και όταν ήρθε ο κύριος Γιούγκερ και μας μίλησε είδαμε ότι δεν λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα όσα ε, απασχόλησαν στις 24 Απριλίου το Συμβούλιο για την ε, διακίνηση των μεταναστών για όλα αυτά τα οποία γίνονται στα χωρικά ύδατα και στα λιμάνια κάποιων συγκεκριμένων χωρών. Στις πρόσφατες διαμοντές με Τουρκία δεν συζητήθηκε το θέμα αυτό, τουλάχιστον ε, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στα ΜΜΕ. Επίσης, ακούμε ότι ασκείται βία κατά χριστιανών είτε στα, στα τόπεδα υποδοχής είτε κατά τη διαδρομή προς την Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για το γίνονται γιατί αυτή η κατάσταση δείχνει πως δεν υπάρχει τελικά εξασφαλισμένη ελευθερία λόγου. Και νομίζω ότι η δίωξη Ιρανών που έχουν προσυλλητιστεί και έχουν γίνει χριστιανοί είναι καλό παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να σιωπούμε ε, μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Δεν μιλώ για μεμονωμένες περιπτώσεις. Άρα, έχω αυτές τις δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' τι γίνεται με την διακίνηση ανθρώπων και την καταπολέμηση του φαινομένου και τι γίνεται με την βία που ασκείται κατά χριστιανών στους καταβλισμούς και στις διαδρομές των μεταναστών. Merci. Euh, moi je trouve... Κύριε Φερζιά, νομίζω ότι συζήτησαμε το θέμα των αλλαγών στις διαδρομές ακούσαμε βέβαια τι έγινε στην Ζάντηση της Βαλέτας και είπαμε ότι τον Απρίλιο ελήφθησαν τα πρώτα μέτρα οπότε και όλοι ε, είχαν κολλήσει στο τι θα γίνει στην Ιταλία και τι θα γίνει με τη διαδρομή Λιβύης Ιταλίας εκεί όπου είχαμε τις βασικές διαδρομές ε, πέρσι όμως τα πράγματα τώρα άλλαξαν, εξελίχθηκαν και οι περισσότεροι περνούν μέσω Τουρκίας Ελλάδος. Και πώς να μην σκεφτεί κανείς ότι η Τουρκία έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε όλα αυτά και δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με τις εξελίξεις στην Συρία. Πώς τα εξηγεί αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει κάνει κάποια ανάλυση της κατάστασης τώρα. Δεύτερο στοιχείο είναι η κατάσταση που αφορά τους ε, πρόσφυγες αφού γίνει η καταγραφή τους. Δεν ξέρω αν σε κάτι και πάνε να καταγραφούν, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και πάρα πολλοί που λένε όχι στην καταγραφή και όλα αυτά τα hot spot, όλα σε αυτές οι επιφυλάξεις των ε, συντρόφων της πολιτικής ομάδας, δίνουν στο να σκεφτούμε ότι έτσι έχουμε κάποια αδικία, κάποια ανισότητα, γιατί έχουμε τους καλούς πρόσφυγες, αυτοί που έχουν από επιλέξιμες χώρες και έχουμε και τους ε, άλλους οι οποίοι θεωρούνται κακοί μετανάστες, κακοί οικονομικοί μετανάστες. Οπότε θα πρέπει να μας διαβιώσετε σε σχέση με όλα αυτά. Κάτι άλλο τώρα, μια διευκρίνηση για τη χρηματοδότηση και για το Ταμείο της ε, Ένταξης ε, το άλλο ταμείο που είπατε δεν, καταλαβαίνω τι γίνεται και τι γίνονται και με αυτά τα καταπιστεύματα τα οποία έχετε προσθέσει σε αυτό το τοπίο 800 ε, εκατομμύρια αλλά τι να σου πω με, με, με, με αυτά τα ποσά που αναφέρετε πως να μην έχουν τόσο νεκρούς στην Μεσόγειο τι γίνεται με τις παραβιάσεις. Εγώ ε, προβληματίζομαι, γιατί και στο καλέ είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις. 20.000. Άλλος. Ο επόμενος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μένουν ένα σωρό απαντήσεις, ε, ε, ερωτήσεις τις οποίες ε, δεν μπορούμε να τις απαιτήσουμε στην Κομισιόν γιατί τελικά δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται τόσε σύνοδοι κορυφή, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Για τους δρόμους των λαθρομεταναστών πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες γιατί οι ετούντες ασύλο έχουν την υποχρέωση να εγγράφονται κατά την είσοδό τους. Τι γίνεται ακριβώς λοιπόν με αυτούς τις οδούς, ε, τι τους ε, ε, δι, τι κάνουμε, αναγνωρίζουμε ακριβώς ποιοι είναι, ποιες είναι αυτές οι οδοί, τους δίνουμε φυλάδια, ξέρουμε πώς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Σχετικά με τα μέτρα μετεκατάστασης, αν πιστέψουμε τον τύπο, ε, έχουν λίγοι μετακατασταθεί σύμφωνα με τα όσα λέει ο τύπος. Ε, τα νούμερα τελικά ε, δεν Ε, σύμφωνα με τον ε, τύπο, 750.000 ε, είναι το σύνολο των μεταναστών, 80.000 θα πρέπει να πάνε στην Γερμανία και άλλοι τόσοι στην Σουηδία. Πραγματικά φτάνουμε σχεδόν στο ένα εκατομμύριο και υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν έχουν τελικά εγγραφεί κατά την είσοδό τους. Τι γίνεται λοιπόν με αυτούς που δεν έχουν εγγραφεί πώς θα εντατικοποιήσουμε την πληροφόρηση για να μπορέσουν να εγγράφονται και ποιες είναι οι κυρώσεις ε, που τελικά θα επιβάλλουμε σε αυτούς που δεν έχουν δηλώσει την είσοδό τους. Αν δεν τα λύσουμε αυτά δεν θα αλλάξει τίποτα. Ευχαριστούμε. Κύριε Φόικτ, ε, έχω και εγώ μία ερώτηση, κυρία Σίγκαν. Η τελευταία συνάντηση για τα Βαλκάνια αποφάσισε να δημιουργηθούν 100.000 θέσεις, για τους μετανάστες. 50.000 στην Ελλάδα, οι υπόλοιποι 50.000 πού θα πάνε. Έχετε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή σας γιατί έχουμε μετά άλλο θέμα. Ευχαριστώ. Για μένα το σημαντικό και η προστιθέμενη αξία είναι να ακούσω τα ερωτήματά σας, αλλά νομίζω ότι χρειάζομαστε στο μέλλον περισσότερο χρόνο για να μπορούμε να συζητάμε σε βάθος τα θέματα αυτά. Αν πρέπει λοιπόν να σας ε, απαντήσω σε 10 λεπτά, θα προτιμούσα να μιλούσε ο συνάδελφος που ήταν εκεί, που μπορούσε να απαντήσει πιο συγκεκριμένα. Είναι κρίσιμη στιγμή, στιγμή αξιοπιστίας για την Ευρώπη, αλλά είναι και μία από τις χειρότερες κρίσεις που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ και όλοι το ξέρουν. Νομίζω ότι το γεγονός ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων συναντιούνται είναι πολύ σημαντικό γιατί μας βοηθά να έχουμε το πολιτικό μήνυμα που θα δοθεί σε όλους μας και μας επιτρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε καλή κατανόηση της κατάστασης. Και ο στόχος μας είναι να κατανοήσουμε καλά το τι συμβαίνει, γιατί όπως είπατε υπάρχουν τόσα δεδομένα, τόσε στατιστικές και τα παίρνουμε και προσπαθούμε να τα δώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και να μπορούμε και εμείς να αντιδρούμε σε πραγματικό χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι όλες αυτές οι πολιτικές αποφάσεις μας δίνουν στην ουσία την εντολή να δουλέψουμε στο πεδίο. Η δουλειά στο πεδίο είναι το πιο σημαντικό που κάνουμε και δεν είναι εύκολη. Ούτε η κατάσταση είναι εύκολη γιατί οι αιτίε της κρίσης είναι εν μέρει εσωτερικές και εν μέρει εξωτερικές. Κάποιες από αυτές δεν εξαρτώνται από μας και υπάρχει μια σωρία πραγμάτων που ε, στην ουσία δεν μας επιτρέπουν την επίλυση της κρίσης. Παίρνουμε λοιπόν κάποιες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για να μπορούμε να δουλέψουμε στο πεδίο και για να προσπαθήσουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Και αυτά τα επόμενα βήματα είναι μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης ε, ημερήσιας διάταξης για τη μετανάστευση, για τη μετεγκατάσταση και τα hot spots είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Τα νομικά ε, ε, εργαλεία που μπορεί να έχουμε, τα νομικά μέσα, το Δουβλίνο που θα αναφέρω σε λίγο, η δουλειά για το Δουβλίνο και η βελτίωση του κοινού συστήματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βοήθεια στην Ελλάδα και συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Αν τα λέω έτσι φαίνονται ότι είναι τα ίδια πράγματα, όμως το περιεχόμενο στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς είναι πολύ απτό και πολύ διαφορετικό σε επίπεδο ποιότητας από το παρελθόν. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Είναι η ευκαιρία μας να χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας αυτή την κατάσταση γιατί όπως είπα και στην αρχική μου ομιλία η ε, οδηγία για τις επιστροφές στις χώρες προέλευσης πρέπει να εφαρμοστεί και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε περίπτωση παραβίασης ε, και τα λοιπά. Και πώς ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο για τις επιστροφές, ε, το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει και επηρεάζει σημαντικά τα ποσοστά επιστροφής. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά σχετίζονται με τις ε, συμφωνίες ε, μεταγκατάστασης και τις συνεργασίες με τις χώρες που θα λάβουν, θα λάβουν μέρος στη διαδικασία εφελούσια ή μη εφελούσια επιστροφής. Έχουμε λοιπόν διάλογο με τις τρίτε χώρες, θα το βρείτε αυτό στα συμπεράσματα της χθεσινής συνάντησης των Υπουργών Εσωτερικών και υπάρχει και διμερής διάλογος σε υψηλό επίπεδο. Συναντήσεις με χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Μαρόκο, η Νιγηρία, το Πακιστάν και η Τουρκία που μας βοηθούν να δούμε ποια είναι τα στοιχεία της επανεισδοχής και της επιστροφής που πρέπει να ενισχυθούν για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και όλα αυτά σχετίζονται πάρα πολύ με τις συμφωνίες επανεισδοχής. Για τα χρήματα τώρα, να επαναλάβω για άλλη μια φορά και μόνο αυτό μπορώ να κάνω, ότι δεν είναι ότι δεν ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα, τα εθνικά προγράμματα προβλέπουν πού πηγαίνουν τα χρήματα σε κάθε κράτος μέλος έχει προβλεφθεί αυτό για τα επόμενα χρόνια. Η έκτακτη ανάγκη όμως ε, είναι εκεί και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Όταν αναφέρατε το Ταμείο της Αφρικής και το πώς θα κάνουμε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε αυτό, νομίζω ότι θα καταλάβουν τα κράτη-μέλη πώς ακριβώς μπορούν να εφαρμοστούν τα project από τους εταίρους στην Αφρική και όταν θα το δουν θα είναι οι πρώτοι που θα ενδιαφερθούν να λύσουν το πρόβλημα επενδύοντας χρήματα, επενδύοντας σε έργα που θα δώσουν πραγματικά αποτελέσματα. Και ε, είναι προς το συμφέρον τους να συνεισφέρουν σε αυτό το, το ίδρυμα. Είναι πολύ σημαντικά το ταμείο, συγγνώμη. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ε, έχουμε στο προσκήνιο μπροστά μας ε, αυτό το έγγραφο, την ανακοίνωση του Οκτωβρίου, αλλά τα δεδομένα καθημερινά αλλάζουν. Στην εισαγωγική μου δήλωση σας είπα ότι αν πρέπει να σας δώσω συγκεκριμένα νούμερα αυτή τη στιγμή, τα νούμερα είναι 105 άτομα που πηγαίνουν στην ε, Σουηδία, ε, Γαλλία και τα λοιπά, ενώ από την Ελλάδα είναι 30 αυτοί που πήγαν στο Λουξεμβούργο. Ε, χρειάζονται λοιπόν ε, πολύ να πολλοί φορείς να συμμετάσχουν, ε, οι συνάδελφοι, γιατί με την κατάσταση θα θυμάστε ότι πριν από καιρό προσπαθήσαμε να κάνουμε τα πρώτα πιλωτικά για τη μετεγκατάσταση. Στους καλούς καιρούς, όταν δεν είχαμε κρίση, θα θυμάστε πολύ καλά στις συναντήσεις μας και στην ε, συναντήσεις με το ΕΑΖΟ πόσο δύσκολο ήταν να εφαρμόσουμε αυτά τα πρώτα πιλωτικά όχι μόνο επειδή τα κράτη-μέλη δεν έδειξαν την αλληλεγγύη που έπρεπε προς τη Μαλτά αλλά γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουν και προβλήματα εφαρμογής. Εκείνη την εποχή χωρίς να έχουμε την οξία φάση της κρίσης κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένε χώρες. Υπήρξε λοιπόν μια πρώτη γεύση για το πόσο δύσκολη είναι η μετεγκατάσταση όμως σε μια κατάσταση κρίσης. Πρέπει να συντάξουμε τις δυνάμει μας και να βοηθήσουμε και βοηθά μάλλον να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές και τη δουλειά στο πεδίο για να μπορούμε να ε, εκτελέσουμε αυτή τη μετεγκατάσταση στην πρώτη αρχική φάση δεν μπορούμε να περιμένουμε να υπάρξει πλήρης εφαρμογή. Αυτό που ήταν σημαντικό σε αυτά που είπα είναι ότι πήραμε μεγάλα μαθήματα, πολύ εμπειρία σε αυτή την πρώτη φάση για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη εφαρμογή. Και κυρία Πρόεδρε, επειδή δεν μπορώ να επισέλθω σε άλλα θέματα, θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία τον επικεφαλή του νομικού τμήματο ε, που πήγε στην Ελλάδα για πέντε λεπτά αυστηρά, λέει η πρόεδρος, ναι, για πέντε λεπτά, να μιλήσει και να μα δώσει απευθείας ε, ε, εικόνα από το τι γίνεται στα hot spots στην Ελλάδα. Και αυτά που θα πει θα απαντήσουν στα σχόλιά σας, αλλά θα είναι και μία άμεση μαρτυρία ενός ανθρώπου που έχει πάει στο παιδεία. Κύριε Σίγκαν παρακαλώ. Κυρία Σπινέλη, να ακούσουμε πρώτα τον κύριο και μετά. Ονομάζομαι Δημήτρης Γιωτάκος, είμαι υπεύθυνο του νομικού Τμήματο της Γενικής Διεύθυνση ε, που εστάλει ε, στην Ελλάδα για να δει πώ ακριβώς ε, γίνεται η προσέγγιση με τα hot spot και την μετακατάσταση των πρώτων ανθρώπων. Δεν θα μιλήσω για την Ιταλία, υπάρχει άλλο ειδικό απεσταλμένο που πήγε εκεί και υπάρχουν πολλές μεγάλες διαφορές και ομοιότητες. Μία μεγάλη διαφορά στην Ελλάδα είναι αυτό που είπε η κυρία Σπινέλη, ότι η χώρα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ε, προβλήματα ρευστότητας, δεν μπορούν να πάνε τα χρήματα εκεί για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες και εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να ε, ε, επέμβει η Κομισιόν. Υπάρχουν διάφορες κοινέ ευθύνε στην Ελλάδα, έπρεπε να αφιερωθεί πολύ χρόνο για να θεσπιστεί το πλαίσιο που θα βοηθήσει στην λήψη των χρημάτων και πολλής χρόνο χάθηκε. Τώρα υπάρχουν οι δομέ, υπάρχουν τα χρήματα, έχουν γίνει ε, κάποιες ε, ε, καταβολές στον κοινό λογαριασμό που έχει ε, η Κομισιόν ε, στην Τράπεζα της Ελλάδος. 33 εκατομμύρια είναι εκεί και περιμένουν να τα χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες το συντομότερο. Όμως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ε, φαίνεται ότι για άλλη μια φορά θα επιληθεί πολύ αργά για τη λειτουργία των hot spot έχω πάει πολλές φορές εκεί. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για αυτά είναι δύο βασικές λειτουργίες. Πρώτον, η εγγραφή, η δήλωση δηλαδή εισόδου που περιλαμβάνει την ταυτοποίηση και τη δακτυλοσκόπηση, τη λήψη των δακτυλικών αποτιμάτων, των υπηκών ε, τρίτων χωρών που φτάνουν στα νησιά και η δεύτερη λειτουργία είναι η στέγαση. Η κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Ένα hot spot υπάρχει στη Λέσβο που είναι σχεδόν πλήρες και υπάρχουν άλλα τέσσερα στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας ε, που είναι υποκατασκευή. Η προθεσμία της ελληνικής κυβέρνησης είναι τέλη Νοεμβρίου. Γενικά η εγγραφή λειτουργεί καλά στην Ελλάδα. Αυτό που λείπει είναι η σωστή και αξιοπρεπή στέγαση γιατί πήγε καλά η δήλωση ε, εισόδου για γεωγραφικούς καθαρά λόγους. Ε, κανένας ε, από τους νεοαφιχθέντες δεν μπορεί να φύγει από τα νησιά και να πάνε αλλού, εκτός αν έχει πλήρως εγγραφή. Υπάρχουν δηλαδή αυστηροί έλεγχοι από την ακτοφυλακή και τη Frontex, από το λιμενικό και τη Frontex, για, στα ferry boat που μεταφέρουν τους ανθρώπους από τα νησιά στην ε, ε, κεντρική Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε μια ειδική συνάντηση ε, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο σημείο νούμερο 7. Ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία λεπτομέρειε συντογή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο. Στην ε, συνάντηση της 10 Η ενδεκάτου πέρσι έγινε μια ανταλλαγή απόψεων. Η κυρία Μέτσολα είναι εδώ αν θέλετε μπορείτε να σου πείτε δύο λόγια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είναι κρίσιμος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το άσυλο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την υπηρεσία αυτή, να τη βοηθήσουμε να πετύχει τους στόχους της. Έχουμε το άρθρο 49 της άσο που ορίζει ότι θα πρέπει να γίνουν σχετικές ρυθμίσεις και έτσι θα πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο για Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λίχτενστάιν οι οποίες θα πρέπει να εμπλακούν στο ε, έργο αυτής της υπηρεσίας. Αυτές οι χώρες θα δώσουν μια καινούργια διάσταση στην ΕΑΣΟ Και έτσι θα υπάρξει συνέχεια στην συλλογή των δεδομένων. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει το πράσινο φως για τη σύναψη συμφωνίας με Νορβηγία και Λίχτενστάιν. Ήδη η Λίμπε έχει εγκρίνει την συμφωνία ε, και το θέμα θα κατέβει για έγκριση στην Ολομέλεια αποφασίστηκε λόγω του δημοσιοφίσματος του Περσίνου στην Ελβετία να αναβληθεί η σχετική συμφωνία. Ανήκει στο σύστημα του Δευλίνου η Ελβετία και συμμετέχει πλήρως. Και όταν γίνει η ρύθμιση ε, των σχέσεων Ελβετίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΔΕΑΣΟ θα έχει ακόμα μια διάσταση και συμφώνησε να συμμετάσχει ε, ε, εκούσια είναι μια δέσμευση που έχει αναλυφθεί και είπαμε ότι έτσι θα έχουμε καταρχήν 1.500 κατόπιν άλλους 1.520 οι οποίοι θα μετεγκατασταθούν. Με το πρόγραμμα αυτό θα αντιμετωπιστεί η μετανάστευση των τελευταίων ετών. κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν γιατί έχουμε την κρίση την προσφυγική που τώρα Οπότε μέχρι τώρα η Ελβετία έχει συμμετάσχει στην πολιτική αυτή ανεπίσημα. Όμως ε, έχει βοηθηθεί έτσι η Ιταλία για ένα σωρό ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από κάποια νομοθετική ρύθμιση. Πάντως, όταν επισημοποιηθεί η σχέση ΕΑΣΟ και Ελβετίας, θα επισημοποιηθεί και η συνεργασία. Οπότε έτσι θα έχουμε βοήθεια από την χώρα αυτή. Και τελικά θα έχουμε μια εναρμόνιση στην πολιτική ασύλου. Σας προτείνω να προχωρήσουμε και να εγκρίνουμε το σχέδιο έκθεσης. Ελπίζω να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι. Έτσι να προχωρήσουμε. Πάντως ε, πριν ε, δευτερολογήσω, ευχαριστώ να ακούσω παρατηρήσεις από τους συναδέλφους. Η κυρία Σιλβικηγιόν που είναι σκιώδης εισηγήτρια. Η Ρομπέρτα μας τα είπε. Οι διαπραγματεύσεις ε, με την Ελβετική Συνομοσπονδία έχουν αρχίσει, αλλά ήταν δύσκολες. Το θέμα αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι συμβολίζει τις αβεβαιότητες που προέκυψαν από το ψήφισμα του Φεβρουαρίου 14. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τα πράγματα ακόμη πολύ σαφώς ως προς τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος του 9 Φεβρουαρίου. Οι συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ Ελβετίας και Ένωσης αφορούσαν κυρίως τα θέματα ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων. Πάνω από 100.000 Ελβετοί συνυπέγραψαν μία πρωτοβουλία για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο σημειώνουμε ότι υπάρχει νομική ασάφεια ως προς το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά βέβαια πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το είπε και η κυρία Μέτσολα, η Ελβετία δέχτηκε να συμμετάσχει εθελοντικά στο πρόγραμμα με την καταστάσεων και συμμετέχει ήδη στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Γραφείου για το Άσυλο, αλλά λείπει ένα επίσημο πλαίσιο και αυτό εμποδίζει τα πράγματα. Η πραγματιστική αυτή προσέγγιση βέβαια δεν αποτελεί εν λευκό επιταγή και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις εξελίξεις γιατί πρέπει να δούμε εάν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος διαφέρει από τις αξίες της Ένωσης. κυρία Βερζιά, ναι, λίγο σαν τη Σιλβίγκη Γιώμ και εγώ, με που βλέπω να ξαναγυρίζει αυτό το θέμα, γιατί ίσως χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τους κοιόδης, για το πότε συζητιούνται τα θέματα, τέλος πάντων. Το θέμα είχε διαγραφεί φύγει από την ημερήσια διάταξή μας μετά το δημοψήφισμα, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα μάλλον. Συμμερίζομαι και εγώ τις αμφιβολίες. Η Ελβετία συμμετέχει στο Δουβλίνο και στο Σέγγεν, στο πρόγραμμα μετεκαταστάσεων και έχουμε την εντύπωση ότι προς στιγμήν, χωρίς να έχει γίνει η μελέτη των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, έχουμε την εντύπωση ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία επιλέγει μόνο ό,τι τη βολεύει. Το ίδιο κάνουν και άλλες χώρες της Ένωσης βέβαια, αλλά αναρωτιέμαι πραγματικά ιδίω για θέματα ασύλου μήπως δεν πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες ως προς το τι πραγματικά θέλουν να κάνουν οι ελβετικές αρχές. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά κύριε Κύρκοπ με τα συγχωρήσεως. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν πρέπει να επικρίνουμε την Ελβετία. Όπως ξέρουμε, η Ελβετία έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε διάφορες διατάξεις ε, και κανονισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως τμήμα των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι θετικό. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μένα, αλλά έχει βοηθήσει την Ένωση για πολλά χρόνια με διαφόρους τρόπους. Δεν θα τους επέκρινα λοιπόν. Νομίζω παρόλα αυτά ότι αν μου επιτρέπετε θα υποστηρίξω κάποιες από τις παρατηρήσεις που μόλις έκαναν οι συνάδελφοι. Η αξία της συνεργασίας είναι πολύ σημαντική, ειδικότερα ε, η συμμετοχή στην ΕΑΣΟ που είναι ένα από τα, ένας από τους οργανισμούς που πρόσφατα στην κρίση που βιώνουμε είχε πολύ θετική συμβολή κατά τη γνώμη μου. Και έχει νόημα ε, η Ελβετία να εμπλακεί στον κανονισμό του Δουβλίνου και στη μακροπρόθεσμη αποτελεσματική εφαρμογή του. Είναι προς το συμφέρον όλων μας αυτό και είναι πολύ θετικό το βήμα όσον με αφορά. Και όσον αφορά στην ομάδα μου, να πω ότι εμείς υποστηρίζουμε πλήρως ε, την θετική αυτή και προσέγγιση της Ελβετίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Βίξτρομ, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ε, ε, μιλάω με, για αυτό το θέμα φέτος ε, ε και η χώρα μου πραγματικά ε, ε, εμπλέκεται τόσο πολύ σε αυτό το θέμα και παρόλο που μιλάω για πρώτη φορά στα Σουηδικά είναι πολύ σημαντικό να το κάνω. Νομίζω ότι είναι το πρόγραμμα αυτό ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί έχει να κάνει με την συνεργασία της Ελβετίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θετικό που μπορεί η Ελβετία να υποστηρίξει την ΕΑΖΟ. Έτσι λοιπόν η ομάδα μου, εγώ ε, και εγώ υποστηρίζουμε πλήρως την κυρία Μετσόλα σε αυτό το θέμα. Σε αυτές τις κρίσιμες μέρες είναι προς το συμφέρον όλων μας να γίνεται κάτι τέτοιο και πρέπει εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε θετικά προδιοτεθειμένοι απέναντι στην Ελβετία. Ε, ας πούμε το γραφείο στη Μάλτα μπορεί και αυτό να συμμετάσχει, να υπάρχει ο διάλογος, όλα αυτά είναι σημαντικά και θετικά. Πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο στο θέμα του ε, ασύλου και της μετανάστασης στην Ευρώπη ε, βλέπουμε συχνά να καταραίει η συνεργασία. Είναι καλό λοιπόν που μια τέτοια χώρα έχει μια θετική συμβολή. Η κυρία Βίξτρομ, η κυρία Μετσόλα ζήτησε το λόγο, αλλά για δύο λεπτά μόνο αν μπορείτε, παρακαλώ. Θα ήθελα, ε, κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους κοιόδες ηγητές που συνεργάστηκαν μαζί μου. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στην προηγούμενη θητεία για τους ευχαριστώ όλους για την ε, υπομονή τους. Κυρία Βεργιά, ξέρετε, κοινοποίησα σε όλους τους ηγητές τη θέση της πολιτικής ομάδας και περίμενα κατόπιν απαντήσεις θετικές ή αρνητικές. Επίσης, έλαβα υπόψη το ότι χρειάζεται να συνεργαστούμε κι άλλο οι εισηγητέ. Ευχαριστούμε κύριε Μέτσολα. Και τώρα έχουμε το επόμενο θέμα το οποίο αφορά ε, το τεχνίδιο αθωότητος και το δικαίωμα παράσταση του κατηγορουμένου στη δίκη. Sur la négociation sur la directive concernant les procédures pénales. Επαναλαμβάνει τον τίτλο της έκθεσης γιατί πρόκειται για μια ε, οδηγία που αφορά την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την ποινική δικονομία σε σχέση με την ερημοδικία και άλλα δικονομικά ζητήματα. Στις 27 Οκτωβρίου έγινε πρώτη συζήτηση, υπήρχε συμφωνία και η Κορεπέρ επιβεβαίωσε 4 Νοεμβρίου και πρόκειται αυτό να ε, συστηθεί στην Επιτροπή μας σήμερα. Θα τώρα το λόγο στην κυρία Ανταλή Γκρισμπέκ που είναι η συγγήτρια. Η κυρία Γκρισμπέκ πρόκειται να μας πει πώς έχει η κατάσταση των ε, διαπραγματεύσεων. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Πέστε μας κυρία Γκρισμπέκ τι συμβαίνει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά να σας πω ότι μετά από πολλούς μήνες προσπάθειας τελικά καταφέραμε να συμφωνήσουμε για αυτήν την οδηγία που αφορά το τεκμήριο της αθότητος. Γιατί κατά τον πέμπτο τριμερή διάλογο στο Στρασβούργο καταφέραμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο και στις 4 Νοεμβρίου η Κορεπέρ ενέκρινε την συμφωνία μας. Να σας πω τώρα τι έγινε με τις διαπραγματεύσεις. Τον Νοέμβριο του 2013 ε, είχαμε τη δέσμη ε, για τα δικονομικά της Βουλής Επιτροπής, το οποίο είχε διάφορες προτάσεις και τα ξέρουμε για το Συμβούλιο Αθωότητος και λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το Συμβούλιο ενέκρινε μια γενική θέση και το Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή μας ε, με τη σειρά της υιοθέτησε κάποιες τελικές θέσεις, οπότε ξεκίνησε γρήγορα ε, ο τριμερής διάλογος τον ε, Απρίλιο, Μάιο και Ιούλιο γίνανε υπό Λετωνική Προεδρία και κατόπιν υπό Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Οπότε ε, σημειώθηκε ταχεία πρόοδος και όσον αφορά την Συμφωνία για το Δημήριο της αθότητας, όσον αφορά την αρχή σύμφωνα με την οποία το πρόσωπο δείξεως το έχει κατηγορούσε αρχή ε, τότε γίνεται αυτό το Συντούμπι προωρέο και υπάρχει ένα καινούριο άρθρο όσον αφορά την, ε, το δικαίωμα παράστασης των κατηγορουμένων ή υπόπτων στην ε, δίκη. Ε, Επίση, υπήρξαν κάποιε διαφωνίε για την αντιστροφή του βάρου αποδείξεω όσον αφορά για το δικαίωμα ενημέρωση, για το δικαίωμα του να σιωπήσει κανεί. Ε, σε σχέση με την ερημοδικία, σε σχέση επίσης με το παραδεκτό των αποθετικών μέσων, οπότε έγινε το Σεπτέμβριο τέταρτος τιμής διάλογος, οπότε και σημειώθηκε αυτή η συμφωνία με το σύνολο των σχεδόν εισηγητών, ε, που του ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή τους και η προσέγγιση τους ε, στάθηκαν αποφασιστικές, ούτως ώστε να φτάσουμε σε τελική πρόταση για να βγούμε από το αδιέξοδο και να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Επίσης, ε, με τρεις προτεραιότητες, την κατάργηση του 5-2 στον φροντίνη τροφή του Βαρσοποδίξεως, που ήταν η πρώτη κόκκινη γραμμή για την ομάδα μας. Τι γίνεται με τις αποδείξεις που αποσπώνται σε παραβίαση του δικαιώματος ε, της ε, σιωπής, επίσης αποδείξεις και ομολογία κατόπιν βασανιστήριων και επίσης το το, το περίφημο άρθρο που είχε σχέση με το και συζητήσαμε την πρότασή μα και καταλήξαμε σε συμφωνία. Αυτά για τα, τα τρία, τους τρεις βασικούς άξονες ε, για το πεδίο εφαρμογή, για το άρθρο 2 είπαμε ότι έχουμε μια, ε, έναν ορισμό ώστε να προστατεύονται οι, οι υποπτοί κατηγορούμενοι. Ε, Από την άλλη μεριά όμως δεν θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία σε νομικά πρόσωπα ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες πράξεις που εμπίπτουν και οπότε δεν θα διέποντα αυτή την ποινική διαδικασία. Αυτό και το άρθρο 4. Επίσης όσον αφορά τη δημόσια ε, ανακοίνωση της ενοχής θέλουμε καλύτερο ορισμό τι θα πει ε, δημόσια ομολογία, τι θα πει δημόσια αρχή, άρθρο 10, τι θα γίνει επομένως σε περίπτωση παραβιάσεως αυτής της αρχής και επίσης αποσπάσαμε μια αιτιολογική παράγραφη όσον αφορά τα μέσα γιατί δεν υπήρχε μια κατηγορηματική ρύθμιση για όσα θέλαμε αλλά τελικά αυτό το οποίο αποσπάσαμε ε, ήταν στα πλαίσια της διαφορετικότητας των ποινικών δικαίων σαν μέλος. Πάντως μπορεί να θεωρηθεί νίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είπαμε ότι υπάρχει τώρα ένα άρθρο το οποίο δεν μπορεί να παρουσιαστεί ε, σε κάποια δίκη, σε κάποια διαδικασία ε, και να περιβάλλεται από στοιχεία που υποδεικνύουν την ενοχή του, ας πούμε χειροπέδες. Επίσης είπαμε ε, ότι για απαλλαγή και για τεκμήριο αυτοδότητας υπάρχουν τώρα άρθρα το 5-2 ήταν τη σοφή κάτω είπαμε ότι αποσπάσαμε μια, την κόκκινη γραμμή αυτό που θέλαμε, 6 και 7 για το δικαίωμα ε, σιωπής. Δεχθήκαμε την κατάργηση του δικαίωματος μη συνεργασία και χάσαμε και την παράγραφο για το δικαίωμα ενημέρωση δυστυχώς γιατί στο Συμβούλιο υπήρχε μια ε, παρεμποδίουσα πλειοψηφία και είχε κάποια επιχειρήματα το Συμβούλιο ότι ήδη υπάρχει κάποια οδηγία που καλύπτει αυτό το σημείο. Ε, επίσης αποσπάσαμε μια ξεκάθαρη ε, παράγραφο για τον εξαναγκασμό και για το δικαίωμα συνεργασίας των υπόπτων. Αυτά μπορείτε να τα θεωρήσετε μια πραγματική νίκη και το δικαίωμα στη σιωπή που είναι απόλυτο δικαίωμα και απαλλαχθήκαμε και από κάποιες ε, διατάξεις ε, που απονεύουν το όπως ε, η παράγραφος που έλεγε ότι το δικαστήριο μπορεί να ερμηνεύσει τη σιωπή κατά του κατηγορουμένου. Το άρθρο 8 για την ερημοδικία δεχθήκαμε αυτό που ήθελε το Συμβούλιο αλλά ξεκαθαρίστηκε το άρθρο 8 ε, παράγραφος 3, την περίπτωση που η εκτέλεση κάποιες απόφασεις ε, για κάποιον ερημοδικούντα είναι δυνατό. Ε, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Επίσης, για τα 11 μέσα έχουμε μια παράγραφο 10, εδάφιο 2, που παραπέμπει στους εθνικούς κανόνες του παραδεκτού των αποδεικτικών μέσων και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα άμυνας και, και, και ε, επίσης στάθμισης των αποδικών μέσων και ένα, μια πολύ καλή σχετική αιτιολογική παράγραφο. Δεν αποσπάσουμε όλα όσα θέλαμε, αλλά και για τα βασανιστήρια επίσης μια διάταξη σημαντική είναι ένα πρώτο βήμα για να υπάρξει ένα ε, ευρωπαϊκό ε, νομοθέτημα μια από όλα αυτά προβλέπονται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί είπαμε ότι αν υπάρχουν βασανιστήρια τότε παραβλέπεται όλη η διαδικασία κοιτάξτε που υπάρχουν επικαλύψεις, 11α καινούργιο άρθρο σε σχέση με τις εκθέσεις ε, και την ενημερώσει ε, της Κομισιόν και το 13 για την επιδιαιτησία ε, και το διάστημα των δύο ετών. Οπότε, Υπάρχει αυτό το νομοθετήμα παρόλα αυτά, όμως έχουμε πάρα πολλές παραβιάσεις ε, σε σχέση με το τεχνείο του αθλητού στην Ευρώπη και για αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτή η συμφωνία και να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε κάποιο χάρτη πορείας για τα δικονομικά δικαιώματα και έτσι η Ευρώπη να σέβεται τα δικαιώματα υπεράσπισης. Εν κατακλείδη ευχαριστώ πάρα πολύ τους και όλους Γιατί με την Κίγκα, την Μπίργκη, την Λόρα, τον Γιάνν, τον ε, Ντένις και τον Κάζι εμείς συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Και να ευχαριστήσουμε και το Συμβούλιο Πρωτοβουλία τη Λετωνική Προεδρία και στη συνέχεια την Λουξεμβουργιανή γιατί κατέβαλαν ε, προσπάθειες ε, προσπάθησαν να, να, να πείσουν να, και επίσης βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. συλλογικά και ομαδικά δούλεψαν. Euh, Ευχαριστώ τώρα δίνω το λόγο σε δύο συναδέλφους μόνο για ένα λεπτό άρα όμως γιατί έχουμε μετά άλλη συνάντηση. Ευχαριστώ η κυρία Γκάλα. Ε, να ευχαριστήσω την Νάταλη Γκρίς. Όλοι ξέρουμε ότι ε, η εισήγηση ήταν ε, ε, παθιασμένη και η δουλειά έγινε με επιμονή ε, μέσα σε δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ήταν όμως η εισηγήτρια εκεί για να αντιμετωπίσει ένα ευαίσθητο θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο όμως διασφαλίζει την αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο την δικονομική διαδικασία. Έτσι λοιπόν, Ε, πετύχαμε όλα αυτά ακριβώς επειδή είχαμε εξαιρετική εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρίσμπεκ. Παρακολούθησα την παρουσίασή της με μεγάλη προσοχή. Ιδιαίτερα την, ε, τις δίκες ερήμην τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συμβιβασμός στον τριμερή διάλογο. Ποιες ήταν οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τις δίκες ερήμην. Άκουσα, είπατε μερικά, αλλά δεν τα κατάλαβα όλα καλά. Άκουσα την αναφορά στο άρθρο 5 ας πούμε. Θέλω να μάθω ακριβώς ποιος συμβιβασμός επιτεύχθη. Ευχαριστούμε κύριε Αγγελάρα. Τώρα μαζί με την Επιτροπή ΑΝΑΦ θα συζητήσουμε. Πετί, πετή. Πετή. Χρήστε κυρά μου. Ευχαριστώ και την Κινγκαγκάλ και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε λέει χρόνο. Θέλετε απάντηση για τις δίκες ερήμην για το 8, όχι για το 5 δηλαδή, γιατί το 5-2 για την αντιστροφή του άχθους της απόδειξης είναι άλλο. Αυτό για το ερήμην ήταν πολύ δύσκολο στη συζήτηση στο Συμβούλιο καταφέραμε οι δίκες ερήμην να μην γίνονται παρά μόνον εάν υπάρχει προσφυγή, εάν έχει πληροφορηθεί ο ενδιαφερόμενος για την δίκη με βάση τέτοιο τρόπο ώστε να πληροφορείται πράγματι, τα κράτη-μέλη δηλαδή να πληροφορούν σωστά γιατί υπάρχουν καταστάσεις όπου ο ύποπτος ή ο καταζητούμενος οργανώνει την φυγή του και επομένως εμείς απαιτούμε τα κράτη-μέλη να πληροφορούν και να μπορεί να γίνει προσφυγή σε δικηγόρο συστηματικά. και να μην υπάρχει δικηγόρος μόνο αν ο ενδιαφερόμενος έχει αποφασίσει να μην πάρει δικηγόρο. Για να βρεθεί έτσι κάποια εξισορρόπηση μεταξύ όσων οργανώνουν φυγή από τη δικαιοσύνη και όσων πραγματικά δεν μπορούν να πληροφορηθούν. Αλλά μπορώ να σας τα πω και άλλη φορά ιδιωτικώς με περισσότερες λεπτομέρειες.